Καθίστε. Να καλωσορίσω τον Μπερμά Κερέ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης για να συζητήσουμε τον ρόλο της ε, ΕΚΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. και βέβαια να συζητήσουμε και τα επόμενα βήματα. Ξέρουμε ότι τη Δευτέρα το Eurogroup αποφάσισε την εκταμείευση ενός, ενός δισεκατομμυρίου μέρους της ε, δόσης που στη συμμόρφωση με τα 15 προαπαιτούμενα. Έχουμε και ένα λοιπόν στο οποίο δεν συνδέεται με τα προαπαιτούμενα, αλλά με την αξιολόγηση της εφαρμογής τη υλοποίηση προηγουμένων μέτρων όσον αφορά την πληρωμή καθυστερημένων οφειλών του ελληνικού δημοσίου και περιμένουμε και αυτό το δεύτερο μέρο τη δόση, Κάτι το οποίο θα επιτρέψει να προχωρήσει και η δεύτερη αξιολόγηση. Διακυβεύονται πολλά σημαντικά ζητήματα, μεταρρύθμιση τη ε, αγορά εργασία, ο προπολογισμό του 2017 κλπ. Και φυσικά έχουμε ανοιχτή ανοιχτό το θέμα της μείωσης του χρέους. Έχουμε τα συμπέρασματα του Eurogroup το Μάιο, πριν το καλοκαίρι. Κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα ήδη αποφασίστηκε να υλοποιηθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, αλλά έχουμε και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ε, μέτρα τα οποία πρέπει να συζητηθούν ε, με την Κομισιόν, με τον ΕΣΕ, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ. Ε, πολύ μπλεγμένη κατάσταση, υπάρχουν πολιτικοί φύσεως περιορισμοί, πολύπλοκες συνθήκες, άλλοι διεθνείς οργανισμοί που εμπλέκονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. θα με ποια μέτρα μέσω πρόθεσμα θα γίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα βεβαίως εδώ μεταξύ, αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι αρκετά. Αυτά είναι τα ζητήματα, κύριε Κουρέ. Έχετε τον λόγο και μετά βεβαίως θα έχετε ευκαιρία να θέσετε ερωτήματα. Κύριε Κουρέ, έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτές. Νομίζω κλέψατε την εισαγωγή μου υπέρ αυτά που ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στην ομάδα εργασία οικονομικής βοήθειας. Κλέψατε όχι μόνο την εισαγωγή μου, αλλά ίσως και κάποιε από τι απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα πω δύο λόγια εισαγωγικός για να σας πω πώς βλέπουμε τον ρόλο της ΕΚΤ στη συζήτηση. Όπως είπα, ευχαριστώ για την ευκαιρία να συμβάλλω στον διάλογο μεταξύ των, ε, της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναφορά αφορά τα προγράμματα προσαρμογής. Και σπίκα, έχει έρθει πολλές φορές εδώ. Έχω έρθει και εγώ, είχα έρθει πριν από δύο χρόνια. Απαντήσαμε σε πολλές και σε πολλές από αυτές τις ερωτήσεις που μας στέλνετε για τα προγράμματα προσαρμογής. Η συζήτηση βεβαίω συνεχίζεται και σήμερα, μια πολύ σημαντική συζήτηση και για μας, καθώς παίζουμε ρόλο στην αξιολόγηση του προγράμματος και την υποπτία. Τα οποία υποπτεύετε και εσεί βεβαίω και η συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα. Μου ζητήσατε να συζητήσουμε κυρίω το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογή στην Ελλάδα από την πλευρά τριπτική γωνία της ΕΚΤ. Τρεις ομάδες παρατηρήσεων έχω για τρία διαφορετικά ζητήματα. Πρώτον, υπενθυμίζω την πολύ δύσκολη κατάσταση πέρσι, το καλοκαίρι του 2015, όταν διαπραγματευόμασταν το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, το τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Με βάση αυτό και αυτό είναι το δεύτερο σημείο, θα μιλήσουμε για το τρίτο πρόγραμμα και τις πρόοδους που έχουν σημειωθεί και βεβαίω τρίτον θα συζητήσουμε τις προκλήσεις για το μέλλον. Χρειάζεται και το υπογραμμίζω και θα το υπογραμμίσω αυτό συλλογική δέσμευση για την επιτυχία του προγράμματο. Να διευκρινίσω επίση ότι στι σημερινέ μου παρατηρήσει θα επικεντρωθώ κυρίω στα οικονομικά ζητήματα, στα χρηματοοικονομικά ζητήματα, γιατί εκεί ε, παίζει ρόλο και αυτά γνωρίζει καλύτερα η ΕΚΤ. Επιθυμίσω λοιπόν τι ε, περιστάσει ε, υπό τι οποίε διαπραγματευθήκαμε το τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Αυτό χρειάζεται αν θέλουμε να καταλάβουμε που βρισκόμαστε σήμερα. Μετά από την βαθιά μακροχρονή ύφεση που ξεκίνησε το 2009, η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας άρχισε να συμβαίνει το δεύτερο μισό του 2014. Μετά όμως από την προκήρυξη εκλογών τέλη Δεκεμβρίου του 2014 άρχισε το κλίμα να επιδεινώνεται ταχύτερα. Η αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική ζωή αλλά και τις εφαρμοσμένες πολιτικές, η αναστροφή μερικών μεταρρυθμίσεων, η απόρριψη δεσμεύσεων από την ε, νέα κυβέρνηση και οι κακές προοπτικές χρηματοδότησης οδήγησαν σε επιδείνωση το οικονομικό κλίμα καθώς και την αξιοπιστία της χώρας, την, χρημα, ε, χρηματοπιστωτική, χρηματοπιστωτική της ε, αξιοπιστία. Μεταξύ του Δεκεμβρίου 14 και του Ιουνίου του 2015 οι εκροές καταθέσεων ανήλθαν σε πάνω από το 1 τέταρτο των συνολικών καταθέσεων αυτό δεν επέτρεψε στην ΕΚΤ να άρει τι απαιτήσει τη όσον αφορά τι ελάχιστε κεφαλαϊκέ απαιτήσει για να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει ω εγγύηση για περαιτέρω δανεισμό. Παρ' όλα αυτά το ευρωσύστημα παρέσχει επαρκή χρηματοδότηση με τη μορφή ρευστότητα στην ελληνική οικονομία για να λειτουργήσει χρήματα τη Κεντρική Τράπεζα από 56 εκατομμύρια ανέβηκε σε 125 δισεκατομμύρια, πάνω από 2 τρίτα του ελληνικού ΑΕΠ. Αυτό νομίζω κάτι παραπάνω από αποδεικνύει την προσήλωσή μα και τη δέσμευσή μα να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία. Νομίζω τα νούμερα μιλούν από μόνα του. Η ρευστότητα, όπω είπα, ε, ανέβηκε που δώσαμε στην Ελλάδα από 56 πάνω από 125 δισεκατομμύρια ευρώ. Τελειουνίου του 2015 περισσότερη βεβαιότητα, ανησυχίε για τις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης ώψη και του προκηρυχθέντο του 5 Ιουλίου 2016. Έκλεισαν οι τράπεζες, εφαρμόστηκαν κεφαλαϊκοί περιορισμοί τέλη Ιουνίου. Αυτό βελτίωσε λίγο την κατάσταση όσον αφορά την ρευστότητα των τραπεζών, αλλά επιδίνωσε τις οικονομικές συνθήκε. Συμφωνήθηκε μετά το τρίτο πρόγραμμα με τι ελληνικέ αρχέ και του εταίρου τη Ευρωζώνη μια προτεραιότητα ήταν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τη αγορά και των καταθετών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Είναι η αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2015 από τον υποπτικό βραχίωνα της ΕΚΤ, τον SSM. Συνεχίσαμε με την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Οι ελλείψεις καλύφθηκαν τα κεφάλαια, αν θέλετε, για την ανακεφαλαίωση καλύφθηκαν κυρίως από τον ιδρυτικό τομέα το δημόσιο περιορίστηκε σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Συμπέρασμα, καταλήξαμε όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα και την ανακεφαλαίωση. Το 2015 είχαμε μια μικρή μείωση του ΑΕΠ, αλλά παρόλα αυτά μία ποσοστή μονάδα καλύτερα από ό,τι περιμένουμε λόγω των κεφαλαϊκών περιορισμών, λόγω των capital controls. Η σταθεροποίηση της ε, παραγωγή ε, οδήγησε σε αύξη, μικρή αύξηση τη κατανάλωση, αύξηση των εξαγωγών και των δημοσίων επενδύσεων. Επιτεύχθη πρωτογενέ πλεόνασμα, χάρη κυρίω σε περιορισμό των δαπανών. Έτσι, ο ελληνικό τραπεζικό τομέα υποφελήθηκε, στήριξε αλλά και υποφελήθηκε από την μακροοικονομική σταθεροποίηση, βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση, αν και δεν ανέκτησε το χαμένο έδαφο ε, αυτό που έχασε δηλαδή, το πρώτο εξάμεινο του 2015. Μετά από την ανακεφαλαίωση τον Οκτώβριο του 2015, ο συνολικό ε, λόγο, το Tier 1, κεφαλαϊκή επάρκεια, δηλαδή το CET1 των ελληνικών τραπεζών, από 11,2 τον Σεπτέμβριο του 2015 ανέβηκε στο 17,9 τον Ιούνιο του 2016. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να φαίνονται πολύ ψηλοί σε, σύγκριση με του μέσου όρου του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματο, αλλά χρειάζονταν οπωσδήποτε χρειάζονταν ένα επιπλέον περιθώριο ασφάλεια για να μπορέσουν οι ελληνικέ τραπέζε να ανταπεξέλθουν στι συνθήκε. Η αποκατάσταση λοιπόν τη κεφαλική επάρκεια των ελληνικών τραπεζών ήταν μόνο ένα βήμα βεβαίω σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρύθμιση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στι ελληνικέ τράπεζε. Τους τελευταίους μήνες εστιάζουμε στα κόκκινα δάνεια και τη διακυβέρνηση των τραπεζών. Η έκθεση σε κόκκινα δάνεια των ελληνικών τραπεζών είναι πολύ υψηλή, 49% τον Ιούνιο του 2016. Ο δεύτερος πληρότερος λόγος, η πόσο το αν θέλετε στην Ευρωζώνη, μετά την Κύπρο, αυτό, η επίλυση του προβλήματος, είναι προϋπόθεση για την παροχή περαιτέρω πιστώσεων χρηματοδότηση στι ελληνικέ τράπεζες και φυσικά για να προκύψει ανάπτυξη. Έγιναν κάποιες νομοθετικές ε, παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Για παράδειγμα, ο νόμος για τα νοικοκυριά επιτρέπει πλέον στις τράπεζες να αντιμετωπίζουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και έτσι καλούνται πλέον οι οφειλέτες δανειολήπτες να πληρώνουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Ο κώδικας δεντολογίας επίσης της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν ένα βήμα. Οι αρχές απελευθέρωσαν τους κανόνες σχετικά με τις απαιτήσει των κόκκινων δανείων. Μπορούν πλέον να πολιθούν με τα δάνεια αυτά και οι τράπεζες έχουν καταστρώσει και συγκεκριμένε στρατηγικέ μέτρα και δράσεις με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητε. Έχουν θέσει δηλαδή συγκεκριμένου αριθμητικούς στόχους για να μειώσουν την έκθεσή του σε κόκκινα δάνεια στο προσεχέ μέλλον. Επίσης, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, έχουμε νέου κανόνε στην Ελλάδα σύμφωνος με τους διεθνείς κανόνες. Η διαδικασία αυτή είναι ακόμα είναι εξελίξη, όμως έχει σημειωθεί πολύ ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά την αναθεώρηση της αλλαγής στα διοικητικά συμβούλια, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι, τα διοικητικά συμβούλια από εδώ και πέρα θα έχουν καλύτερη γνώση, περισσότερη πείρα και ανεξαρτησία. Αυτά πολύ συνοπτικά. Εξελίξεις που άρχισαν να αποφέρουν και κάποια αποτελέσματα. Έτσι η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται πλην όμως με αργό ρυθμό. Οι τράπεζες μπορούν να δανειστούν από την αγορά με υψηλής ποιότητας εγγυήσεις και η, ως προς την ρευστότητα μειώθηκε η εξάρτηση από την Κεντρική Τράπεζα από την ΕΚΤ στα 78 δισεκατομμύρια, κάτω από τα 125 που έλεγα λίγο πριν. Η πρώτη λοιπόν αξιολόγηση είναι ένα πρώτο βήμα για περισσότερη σταθερότητα. Ετοιμάζουμε το έδαφος για ανάκαμψη της οικονομίας και έξοδος της αγορές. Όμως, μένει πολλή δουλειά μπροστά μας. Το γεγονός ότι οι καταθέσει τη τράπεζα είναι ακόμη στα 3 τέταρτα των επιπέδων του τέλου του 2014, δείχνει πόσο μεγάλε είναι οι προκλήσει. Και όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο εάν εφαρμοστούν αυτέ οι πολιτικέ και υποστηριχθούν πολιτικά από όλου του εμπλεκομένου Από χρηματοοικονομική άποψη να τονίσω δύο προαπαιτούμενα για την επόμενη αξιολόγηση που είναι κινήσει οι οποίε θα διευκολύνουν την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Αυτό είναι το πρώτο που είπα. Προ τούτο χρειάζεται πρώτον η δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης αυτών των ε, δανείων. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για πιστωτές και οφειλέτες να συνεργαστούν στο πλαίσιο αυτό. Και το δεύτερο προαπαιτούμενο είναι η ανάπτυξη του κώδικα του πτωχευτικού κώδικα για να αναδιαρθρωθεί και ο μη χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα. Πέρα από αυτέ τι νομοθετικέ πρωτοβουλίε, οι ελληνικέ αρχέ πρέπει να εφαρμόσουν τα συμπεφωνημένα μέτρα για να βελτιώσουν τη δικαιοσύνη, να επιταχυνθεί η διεξαγωγή των δικών και να ισχυροποιηθούν τα δικαστήρια, οι διοικητικέ του ικανότητε. Αυτά δεν είναι μόνο ελληνικά προβλήματα. Στην Ευρωζώνη γενικότερα ξέρουμε ότι το θέμα των κόκκινων δανείων απαιτεί περισσότερη νομοθέτηση. Βέβαια στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Αυτέ οι μεταρρυθμίσει απαιτούνται για την υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, δράση χρειάζεται στου τρει αυτού πυλώνε, όπω προείπα. Πρώτον, να βελτιώσουμε την δημοσιονομική θέση τη Ελλάδα. Δεύτερον, να αποκατασταθεί βιώσιμη ανάπτυξη με μεταρρυθμίσει. Και τρίτον, να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο κράτο, σύγχρονη διοίκηση και ένα σύστημα κοινωνική ασφάλιση με συγκεκριμένου στόχου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογή αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν σοβαρέ προκλήσει που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου. Η ΕΚΤ, γνωρίζεται έχει υποστηρίξει μια ανάλυση βιωσιμότητας, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρέ ανησυχίε όσον αφορά, σοβαρέ αμφιβολίε όσον αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου. Όπω γνωρίζετε, στο Eurogroup συνεχίζεται η συζήτηση για τα πρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ε, για να δούμε πώ θα εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου. Προσβλέπουμε σε λύση η οποία θα διαβεβαιώσει τι αγορέ, η οποία θα αποκραστεί στην εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα του χρέου. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή του ΔΝΤ και βεβαίω να δώσουμε την προοπτική στην Ελλάδα να βγει στι αγορέ μετά το τέλο του προγράμματο ή και πριν το τέλο του προγράμματο, τον Ιούλιο του 2018. Και φυσικά πρέπει να υποστηρίξουμε τι μεταρρυθμίσει για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να βγει η Ελλάδα στι αγορέ με διάρκεια και βιωσιμότητα. Πρέπει οι ελληνικέ αρχέ να παραμείνουν προσιλωμένε στου στόχου και τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματο. Μόνο αν συμβεί αυτό, τότε όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έχουν την βεβαιότητα ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα γυρίσουν προς τα πίσω, αντιθέτως θα ενισχυθούν με... και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Συμπερασματικά λοιπόν, σας είπα τι έχει γίνει ως σήμερα, σας είπα ποιες είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα εν του τρίτου και κατά τη διάρκεια του τρίτου προγράμματο προσαρμογή, οι Ευρωπαίοι ηγέτε συμφώνησαν μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν το μέλλον και την παραμονή τη Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ. Και βεβαίω εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί στην, της έκτος όσον αφορά το, την χρηματοδότηση της χώρας. Αν ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει, είμαι πεπισμένος ότι στο τέλος η Ελλάδα θα μπορέσει να υποφεληθεί από τα ωφέλη της ε, Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης της ναι. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να γίνει ισχυρότερη σε μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Πάντως η Ευρώπη, να ξέρετε, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τι πιέσει ασφάλεια και μετανάστευση χωρί μια ισχυρή και βιώσιμη οικονομία. Και αυτό ε, προποθέτει μια ισχυρότερη ΟΝΕ. Ναι. Φυσικά και εδώ η Ελλάδα έχει πολλή δουλειά μπροστά τη. Η έκτατη μεριά τη θα κάνει την πορεία να βελτιώσει το και να ενισχύσει το πλαίσιο. Εμείς ως Κεντρική Τράπεζα της Ευρωζώνης, αλλά και η, Ευρωπαϊκή, και η Ελληνική Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, θα κάνουν ε, ό,τι μπορούν προς την κατεύθυνση αυτή. Είμαι έτοιμος να ακούσω ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Βεβαίως ε, υπάρχουν πολλά βασικά παραδοτέα από όλους μας για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ο κύριος Κύρτσος είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιες θετικές και κάποιες αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ε, ε, ε, ήθελα να ρωτήσω αν οι ειδικοί έχουν αναλύσει την κατάσταση της τράπεζας. Καταρχήν, ε, έχουμε ε, αύξηση των φορολογικών εσόδων ε, από το Σεπτέμβρη και αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τα προηγούμενα δύο χρόνια γιατί είχαμε αύξηση φόρων αλλά χωρίς αύξηση των φορολογικών εσόδων. Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ υπάρχει μια πολύ ικανοποιητική σε μηνιαία βάση αύξηση των φορολογικών εσόδων. Πιστεύετε ότι αυτό, αν το έχετε αναλύσει, θα συνεχιστεί Υπάρχουν και δύο αρνητικές εξελίξεις. Οι εξαγωγές μειώνονται το 2016 και αυτό είναι περίεργο με την έννοια ότι μειώθηκε το κόστος εργασίας και θεωρητικά θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Οπότε πώς εξηγείται αυτό το πράγμα. Επίσης, τα έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν μειώνονται, γιατί συνεχίζεται η διαδικασία, κατά 3-4% παρά το γεγονός ότι είχαμε ρεκόρ αριθμό τουριστών επισκεπτών στην Ελλάδα. Ε, είναι πιο ανταγωνιστικές οι τιμές, υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχουν ε, προβλήματα, αλλά δεν ξέρω μια απάντηση σε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ για, την, για τις ερωτήσεις. Για τα φορολογικά έσοδα, οι τελευταίες εξελίξεις είναι θετικές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την εταιρική φορολόγηση. Αντιλαμβάνεστε ότι από πλευρά θεσμών θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πάντοτε. Δεν ξέρουμε πόσα μπορούν να ε, μεταφερθούν ε, ε, από το 16 και αν θα συνεχιστούν το 17 Προσοχή λοιπόν ε, για να καταλάβουμε το επακριβές αίτιο της αύξησης των εσόδων από τους φόρους. Δεν θα ε, βασιζόμουν πάρα πολύ σε αυτό το στοιχείο. Θα ήθελα περισσότερα στοιχεία. Για τον τουρισμό ε, δεν τα ξέρει αυτά τα θέματα η ΕΚΤ, όπως αντιλαμβάνεστε. Από πάντως βεβαίως είναι σημαντικό κομμάτι του ελληνικού ΑΕΠ, πρέπει να το δούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε μια μετάθεση ε, στην ε, ε, εξέλιξη των τουριστών, προέλευση κλπ. υπάρχει και γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια, βεβαιότητα στην περιοχή ε, πολλοί ε, τουρίστες ε, φοβούνται να πάνε σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Αν δηλαδή προέρχεται από γειτονικέ χώρες ο τουρισμός, τότε τα έσοδα πέφτουν. Δηλαδή πρέπει να δούμε και, τη, όπως σας είπα, την προέλευση των τουριστών. Αλλά δεν είναι αυτό το βασικό μας αντικείμενο. Ο κύριος Μπούλμαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε κύριε Κορέ. Όταν επισκεφθήκατε ως ε, αντιπροσωπεία αυτής της ομάδας εργασίας τεχνικής, ε, οικονομικής στήριξης στην Ελλάδα, κάνατε συζητήσεις και ε, με συναδέλφους στην Εθνική Κεντρική Τράπεζα και η εικόνα ήταν ότι μας είπαν οι ε, εκπρόσωποι της τράπεζας ότι γενικά αν δείτε τις πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης ε, είναι ε, προσανατολισμένη προς ε, υγιείς οικονομικές σχέσεις. Είναι πολύ περισσότερο αισιόδοξα τα πράγματα τώρα. Αυτά μας είπαν από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα όταν επισκεφθήκαμε τη χώρα ως ομάδα εργασίας οικονομικής στήριξης. Εσείς ημερίζεστε αυτήν την εικόνα. Δεύτερον, υπάρχουν φήμες ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να τεστάρει την κατάσταση στις χρηματοοικονομικές αγορές, στις κεφαλαίες τον επόμενο χρόνο. Ε, τι θεωρείτε, αν γίνει αυτό, ότι θα ε, είναι οι ε, πραγματικές συνθήκες για κάτι τέτοιο. Επίσης υπάρχει, οι Λατίνοι έλεγαν «pacta sunt servanda». Αν υπήρξε συμφωνία μεταξύ ηγετών για πραγματικές μεταρρυθμίσεις και πραγματική ελάφρυνση χρέους από την άλλη, δεν είναι τώρα ώρα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και να βάλουμε και αυτό το θέμα επιτάπητος. Σύνδεση μεταρρυθμίσεων με ελάφρυνση του χρέους λοιπόν. Ευχαριστώ για την αλλαγή στο κλίμα. Υπάρχουν ε, θετικές εξελίξεις από την Ελλάδα όπως περιέγραψε και η Τράπεζα της Ελλάδος. Θα συμφωνούσα ότι η ό,τι αφορά την ε, ποιότητα συνεργασίας μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και των τεσσάρων θεσμών και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το καλοκαίρι του 2015. Οι συζητήσεις με τους Έλληνες ομολόγους είναι πάρα πολύ φιλικές και επικοδομητικές Βεβαίω, ε, βεβαίως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, ε, σοβαρές συζητήσεις, ε, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά το πλαίσιο για τις συζητήσεις τώρα είναι ευεπίφορο και θα οδηγήσει σε πρόοδο, πράγμα που δεν συνέβαινε για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το καλοκαίρι του 2015. Και θέλω μάλιστα να συγχαρώ ιδιαίτερα τον ε, Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος έπαιξε προσωπικά πολύ χρήσιμο ρόλο, δημιουργώντας αυτές τις ε, σχέσεις εργασίας. Υπάρχουν αλλαγές λοιπόν στις μεθόδους εργασίας και πάω τώρα και στα αποτελέσματα. Ε, είχαμε πολλές απογοητεύσεις και προβλήματα στις προβλέψεις με την Ελλάδα, για την Ελλάδα από το 10 μέχρι το 14. Είχαμε πολλές συνεχείς απογοητεύσεις γιατί και οι προβλέψεις μας ήταν πολύ αισιόδοξε σε σχέση με τα αποτελέσματα. Για πρώτη φορά όμως το 2015 και μέχρι τώρα το 2016 υπάρχουν θετικές εξελίξεις και εκπλήξεις σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ ειδικότερα. Λοιπόν, έχουμε θετικές και σε εκπλήξεις και θετικότερο κλίμα λοιπόν. Όταν πρόκειται για την πρόσβαση στις αγορές, όταν μιλάμε γι' αυτό, σίγουρα αυτή η απόφαση θα ληφθεί από τον Υπουργό των Οικονομικών και οι ελληνικές αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν και θα κρίνουν πότε έχει νόημα να βγουν στις αγορές ένα προσωπικό σχόλιο με βάση την προσωπική μου πείρα ως διαχειριστής δημόσιου χρέους, γιατί αυτό ήταν η δουλειά μου, έχει νόημα να τεστάρουμε τις αγορές σταδιακά, αλλά ειλικρινά δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά από αυτή τη διαδικασία, εις ό,τι αφορά δηλαδή την ελάφρυνση των χρηματοδοτικών αναγκών για τον επόμενο χρόνο. Θα υπάρξει μια αλληλεπίδραση με τους επενδυτές και τις αγορές για να δούμε ε, τι επίπτωση θα έχει στο χρέο. Δεν θα είναι μεγάλη επίπτωση, αλλά νομίζω ότι αν μπορεί κανεί να βγει στι αγορέ, αυτό είναι θετικό. Τέλο, ει ό,τι αφορά την ερώτηση για το Πάκτα Σερβάντα, όπω είπα στην εισαγωγή μου, υπάρχουν δεσμεύσει από όλε τι πλευρέ και οι δεσμεύσει θα πρέπει να τηρηθούν και να εκπληρωθούν από όλε τι πλευρέ και υπάρχει σαφή δέσμευση ε, να αντιμετωπιστεί το θέμα του, της βιωσιμότητας του χρέους και εμείς είχαμε εκφράσει σοβαρές ε, επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και αυτό έχει σχέση με την προηγου, τις προηγούμενες ερωτήσεις. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρχει ε, σοβαρή, ε, σοβαρό άνοιγμα στις αγορές χωρίς να είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Όλα είναι αλληλένδετα και συνειφασμένα. Ναι, λοιπόν, ε, η συζήτηση ε, θα, πρέπει να κάνει τη, θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση για το χρέος. Τώρα βεβαίως ο ESM είναι εκείνο που ε, δίνει το στίγμα. Είμαστε σε μια τεχνική φάση όπου αξιολογούμε διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση του χρέους και κυρίως ο ESM είναι εκείνο ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει μέτρα βράχη πρόθεσμα για το χρέος. Ο ESM λοιπόν θα, το, θα πρέπει να τα δει όλα αυτά. Τώρα υπάρχει μια σειρά και η προϋπόθεση για να είναι ε, καλή η συζήτηση θα είναι ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα, στις απαιτήσεις του προγράμματος η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι προφανές. Όλα εξαρτώνται από την ε, ε, αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Κερέ, θα μιλήσω στα ελληνικά. Θα χρειάζεται. Υπάρχει μετάφραση διερμηνία από τα ελληνικά. Η, ερωτήση, η πρώτη ερώτηση μου αφορά την, ε, τα μη εξυπηρετούμενα... Yeah. Number seven, I ε, Η πρώτη ερώτηση μου αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα NPLs. Επειδή αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πραγματικά ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, 40% του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας και έχουμε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανέργους. και οι προσφορές που προτίθεται να κάνουν τα distress funds για να αγοράσουν τα στεγαστικά δάνεια είναι της τάξης του 20% περίπου. Η πρόταση που είχα διαμορφώσει από τον Ιούνιο στη αντίστοιχη συζήτηση που κάναμε στην Αθήνα είναι πρώτα απ' όλα να δοθεί το δικαίωμα πρώτης προσφοράς στο δανειολήπτη ή στον εγγυητή. Αν έχει αυτό το 20% του ποσού να αγοράσει το στεγαστικό του δάνειο. Και αυτό να είναι υποχρέωση εκ μέρους των τραπεζών να απευθυνθούν πρώτα στους ίδιους τους δανειολήπτες. Και το δεύτερο, επειδή μπορεί οι δανειολήπτες να μην έχουν ούτε αυτά τα χρήματα, να φτιαχτεί ένα δημόσιο ταμείο όπως είχε προτείνει ο κύριος Δράγκη και για την Ιταλία. Και σε αυτό το δημόσιο ταμείο να μπορούν να προσφεύγουν οι δανειολήπτες προκειμένου να πάρουν χρήματα για να πληρώσουν το ποσοστό που πρέπει να πληρώσουν για να αγοράσουν το δάνειό τους. Τα χρήματα αυτά μπορούν να βρεθούν διότι έχουν περισσέψει 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το τρίτο δανειακό πακέτο. 25 δισευρώ ευρώ ήταν να πάνε για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, χρησιμοποιήθηκαν μόνο 5,5 επομένως περίσσεψαν 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα θα μπορούσαν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ να πάνε σε αυτό το δημόσιο ταμείο και έτσι οι δανειολήπτες να μπορούν να παίρνουν μια οικονομική ενίσχυση, ένα δάνειο από αυτό το ταμείο, για να μπορούν οι ίδιοι να ξεπληρώσουν το δάνειό τους, αντί να το πάρουν τα κοράκια στο 20%. Και σε αυτό θα ήθελα να έχω την άποψη της ECB, γιατί εσείς είστε ο οργανισμός που παρακολουθεί το θέμα της ε, λειτουργίας των κόκκινων δανείων. Και το δεύτερο, η δεύτερη ερώτηση αφορά την ρύθμιση του χρέους της Ελλάδος. Γιατί δεν χρησιμοποιείτε εσείς, να προτείνετε ο CCB, το μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το IMF για την Ουκρανία. Στην Ουκρανία λέτε ότι θα πρέπει να γίνει, σε σχέση με τη ρύθμιση του χρέους της Ουκρανίας, ένα haircut της τάξης του 20% και εξόφληση του δανείου της Ουκρανίας με ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή αν έχει ανάπτυξη η χώρα να σας πληρώνει. Αν γίνει αυτή η ρύθμιση σημαίνει για την Ελλάδα τουλάχιστον για του χρόνου μία διευκόλυνση της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Διότι θα πληρώσει ένα 0,7% ουσιαστικό η Ελλάδα, λόγω ανάπτυξη, αν έχει του χρόνου, και έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα διευκόλυνση. Γιατί δεν δέχεστε αυτό το μοντέλο της Ουκρανίας, αντί να έχουμε αυτό που κάνουμε σήμερα στην Ελλάδα, που για να εξοφληθούν τα χρέη την επόμενη χρονιά θα πληρώσουμε 8 δισεκατομμύρια ευρώ, με 8,5. Σα ευχαριστώ. Okay, thank you for your, for your Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Για... Θα αρχίσω με τη δεύτερη που αναφέρθηκατε στην Ουκρανία. Η ΕΚΤ, για να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν αποτελεί άμεσο συζητητή για το χρέος, δεν είναι δικά μας τα λεφτά, μπορούμε να δώσουμε συμβουλές για τη βιωσιμότητα, το κάναμε και στο παρελθόν, το κάνουμε και στο μέλλον, Ονομοδοτούμε σχετικά με το τι είναι καλό για τη μεγιστοποίηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των αγορών, αλλά δεν μπαίνουμε στις διαπραγματεύσεις για το χρέος. Αυτό επαφίεται στα κράτη-μέλη, στα πλαίσια του ESM. Η άμεση μου αντίδραση θα ήταν ότι δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, γιατί είναι διαφορετικές οι χρηματοοικονομικές ε, ρυθμίσεις. Ε, η Ουκρανία εξαρτάται κυρίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ η Ελλάδα εξαρτάται από τη χρηματοδότηση του ESM με διαφορετικές προϋποθέσεις. Του ESM η χρηματοδότηση είναι, έχει πολύ πιο πολλές παραχωρήσεις ε, ε, και σε ό,τι αφορά τα επιτόκια και τις περιόδους χάριτος είναι πολύ πιο ευνοϊκές. Το πλαίσιο είναι διαφορετικό λοιπόν και αυτή είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει ε, στο ESM, στο Συμβούλιο του ESM ή στην Ευρωζώνη. Ε, πάντως, πάντα πάνω στη βάση του ESM. Είπα πιο πριν ότι εμείς στην ΕΚΤ πιστεύουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να μετέχει και μετέχει ουσιαστικά, πρακτικά, συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσεις. Ε, δεν υπάρχει συμφωνία για ε, αξιολόγηση χωρίς συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χρειάζεται μεταξύ άλλων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί μπορεί να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ε, διεθνώς. Ε, θα εφαρμοστεί η ίδια μεθοδολογία και τα κριτήρια για την Ελλάδα όπως εφαρμόζουν, ε, εφαρμόζουν και οι άλλες χώρες. Και αυτό είναι μια ε, διασφάλιση, μια εγγύηση απέναντι ε, ως προς το ενδεχόμενο ειδική μεταχείριση της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτός, σε αυτό συμβάλλει το δούνο του Τώρα, για την πρώτη ερώτηση, την προστασία δηλαδή των ιδιοκτητών και των οικοκυριών, αυτό απετέλεσε κομμάτι της συζήτησης, ιδιαίτερα στην πρώτη αξιολόγηση, και συμφωνήσαμε ως θεσμοί και το Eurogroup συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρχει κάποια προστασία για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Θα πρέπει να είναι περιορισμένη και προσωρινή η προστασία αυτή, διότι δεν ξεχνάμε το βασικό στόχο, τον πρωταρχικό στόχο της μεταρρύθμισης της αγοράς. Ε, ε, ο στόχος, εις ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια και τα πτωχευμένα νοικοκυριά, είναι να ε, υπάρξουν ε, ομόλογα που να μην είναι επιβαρημένα με κόκκινα δάνεια. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ε, αυξηθεί η ε, δανειοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Προστασία λοιπόν ναι για τα νοικοκυριά, αυτή όμως μπορεί να δοθεί και μέσω άλλων μέσων. Και εμεί επιμέναμε ε, πολύ να δημιουργηθεί ε, ένα πρόγραμμα γενικού βασικού ε, εισοδήματος, ε, ελάχιστου εισοδήματος. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει για να προστατευτούν τα ευάλωτα νοικοκυριά και, ε, γιατί αν γίνει μέσα του, μέσα του κανονισμού για τα κόκκινα δάνεια θα δημιουργήσει στρεβλώσεις ε, και ανεπιθύμητες ε, επιπτώσεις γιατί δημιουργεί υπερβολικά βάρη και είναι πολύ δύσκολο να δοθούν νέα δάνεια στην Ελλάδα έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσει και όπως γνωρίζετε υπάρχουν δύο διαφορετικές προστασίες για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Υπάρχει ένα πρώτο επίπεδο προστασίας, είναι ο αναθεωρημένος νόμος Κατσέλη όπου αν τα νοικοκυριά είναι κάτω από ένα ε, επίπεδο εισοδημάτων, ε, νομίζω 1,7 ε, επί τα κόστος διαβίωσης και εξαρτάται από το μέγεθος του νοικοκυριού, αν είναι κάτω από ένα όριο ετήσιου εισοδήματος, τότε μπορεί να ε, παρέμβει η κυβέρνηση. Έχει γίνει δεκτό από το πρόγραμμα η, ε, η οικονομική, δημοσιονομική ικανότητα να χρησιμοποιηθεί για να προστατευτούν αυτά τα ε, νοικοκυριά. Και με τον καινούριο νόμο υπάρχει προσωρινή εξαίρεση ε, για όλες τις πρώτες κατοικίες κάτω με αξίας κάτω από 140.000 ευρώ το, το 16-17. Για δύο χρόνια δηλαδή υπάρχει αποτελεσματική προστασία των πιο ευάλωτων ε, νοικοκυριών που είναι πολλά τα νοικοκυριά αυτά τα οποία έχουν ε, κατοικίες αξίας κάτω από 140.000 ευρώ. Είναι μεγάλος λοιπόν ο Αριθμό των οικοκυριών που δεν εμπίπτουν στο νέο αυτό πρόγραμμα. Η Σιλβί Γκουλά. Ευχαριστώ που ήρθατε. Θα μιλήσω γαλλικά. Με ενδιαφέρει το εξή και ευχαριστώ για όλε τι πληροφορίε που μα δώσατε. Τι γίνεται στην πράξη, τόπου. δηλαδή, επαληθεύετε την υλοποίηση, μετράτε τη φτώχεια, Ποια είναι τα συμπεράσματά σας επαναστοχεύετε τις πολιτικές σας, τις αναπροσαρμόζετε και τι θα γίνει στο μέλλον. Και δεν ρωτάω μόνο για την Ελλάδα. Γιατί πραγματικά είμαι απογοητευμένη από τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Έχουμε και το δημογραφικό πρόβλημα τι γίνεται, πού πηγαίνουμε μακροπρόθεσμα και τι γίνεται με την πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Θα μιλήσω και εγώ, θα απαντήσω και εγώ στα γαλλικά. Για το δεύτερο τμήμα της ερωτήσής σας υπάρχει σύνδεση βεβαίως Ελλάδας και υπόλοιπης Ευρωζώνης. Από τη μια μεριά χαιρόμαστε που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι υπουργοί οικονομικών έλαβαν αποφάσει για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι καλό και αποδεικνύει ότι η, Ευρώπη, η Ελλάδα με συγχωρείτε παραμένει αναπόσπαστα δεμένη στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι, το ένα. Όμω δεν υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα, αυτό είναι το ένα, και πολύ χαμηλή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνιστικότητα, είναι και το θέμα χαμηλή ζήτηση στην Ευρωζώνη γενικώ. Όλες οι πρωτοβουλίες για την αναθέρμανση της ζήτησης στην Ευρωζώνη ωφελούν και την Ελλάδα βεβαίω και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ό,τι γίνεται για την Ευρωζώνη είναι καλό και για την Ελλάδα. Οπότε η ΕΚΤ κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ότι της επιτρέπει η εντολή της στο πλαίσιο της νομισματικής της πολιτικής για την ανάπτυξη αυτά σε πρόθεσμη βάση. Το μακροπρόθεσμο είναι άλλον ιστορία. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για την Ελλάδα. Πώ το μετρούμε τώρα, πώ μετρούμε την απόδοση των πολιτικών επιτόπου. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο διότι το πρόγραμμα είναι μακροοικονομικό. Και είναι κίνδυνος, υπάρχει όντω ο κίνδυνος να συνεχίσουμε να μιλάμε μόνο για τα μακροοικονομικά χωρί να βλέπουμε τι γίνεται στην πράξη, στην αγορά. Έχω την αίσθηση ότι μαθαίνουμε, μαθαίνουμε από την αρχή του προγράμματος προσαρμογή το 2010 και σταδιακά συνεργαζόμαστε όλο και περισσότερο με τους άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Από θεσμικής ε, απόψεως τουλάχιστον, η Παγκόσμια Τράπεζα, για παράδειγμα, συμμετέχει στα κοινωνικά θέματα, στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, για παράδειγμα, και την γενίκευση του μέτρου σε όλη τη χώρα, την επέκταση του ελάχιστου εγγυημένου εισόδηματος σε όλη τη χώρα, θα είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για την ελληνική κοινωνία και υπάρχει βέβαια και το φορολογικό, το ασφαλιστικό, αν και από εκεί θα πρέπει να είχαμε ξεκινήσει. Και δεν λέω ότι φτάνει εδώ οι θεσμοί, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, η Κομισιόν και η ΕΚΤ ε, είχαν, πει, είχαν ζητήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα παλιότερα. Ε, αυτή τη στιγμή υλοποιείται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Εν πάση περιπτώσει, το λέω για να πω ότι και η Παγκόσμια Τράπεζα συμμετέχει στην προσπάθεια, αλλά και στη γενικότερη συζήτηση. Όλα αυτά θα αποτελέσουν και αντικείμενο της δεύτερης αξιολόγησης. Και από εκεί και πέρα θα χρειαστούμε μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα αξιολογήσει κατά πόσον το έργο των ελληνικών αρχών είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και πρότυπα. Και δεν θα τελειώσουμε το καν εκεί. Έτσι. Οι εμπειρογνώμονε εξάλλου δεν συμφωνούν αναγκαστικά μεταξύ του. Και μετά θα περάσουμε στην πολιτική συζήτηση σε επίπεδο Eurogroup. Πάντως, θα ζητήσουμε πρώτον τη γνώμη ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, να έχουμε μια τεχνική βάση συζήτηση και για να πω και κάτι για το μέλλον, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τι αξιολογήσει, να αξιολογήσουμε τα πάντα, μόνο για την τρέχουσα αξιολόγηση, για να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με το πώ θα βελτιώσουμε την προσέγγιση μα και πώ στο μέλλον θα βοηθούμε τι χώρε που έχουν ανάγκη. Ξέρουμε ότι ο σημερινό μηχανισμό δημιουργήθηκε εκ των ενόντων το 10. Είναι ατελή βεβαίω, όπω είναι ατελή και η ΟΝΕ. Είναι ο μηχανισμό αν θέλετε, της Τρόικας. Με αυτό δουλεύουμε σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν ένα μονιμότερος μηχανισμό. Πρέπει να γίνουν οι παρετές θεσμικές ρυθμίσει. Αυτό παίρνει χρόνο. Θέλει και μια πολιτική απόφαση. Η ΕΚΤΑ θα πάρει και αυτή τις αποφάσεις τη, αλλά πολύ περισσότερο χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις σε υψηλότερο επίπεδο για όλα τα προγράμματα στην Ευρωζώνη. Χρειάζεται όμω μια επιπλέον διάσταση. Το είπατε και εσείς νομίζω. Το θέμα είναι πώς στη συζήτηση για τα προγράμματα θα σωματώσουμε τη γνώση από την αγορά, από την πραγματικότητα την ίδια και πρέπει να ενσωματώσουμε βεβαίω και την κοινωνική προστασία. Την τελευταία φορά που ήμουν εδώ και συζητούσαμε πριν από δύο χρόνια, είχα κατακλείδη πει ότι ένα από τα προβλήματα που είχαμε στην Ευρωζώνη είναι ότι έχουμε ε, προγράμματα χωρί την Παγκόσμια Τράπεζα. Δηλαδή είχαμε δονητού χωρί την Παγκόσμια Τράπεζα. Το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ όπου πηγαίνει, πηγαίνει με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Τράπεζα Περιφερειακής ανάπτυξη για την ε, μικροοικονομική υποστήριξη, αν θέλετε, των προγραμμάτων και για την παροχή και κοινωνικής προστασίας. Εδώ κινηθήκαμε με βάση τα διαρθρωτικά ταμεία, υπάρχει το Ταμείο Συνεχής. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να γίνει ανακατανομή πόρων. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε τι κάνει ο κάθε θεσμό, ποιοι θεσμοί πρέπει να εμπλακούν, τι είδου δημοσιονομικά εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε για την κοινωνική προστασία κατά τη διάρκεια τη προσαρμογή. Αυτά έχουμε μπροστά μας. παρακαλώ να είμαστε όλοι λίγο πιο σύντομοι, γιατί αρχίσαμε βέβαια με καθυστέρηση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης. Καλώς ήρθατε κύριε Κερέ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας, γιατί θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα τα ελληνικά. Κύριε Κερέ, μας δώσατε χρήσιμες και αισιόδοξε πληροφορίες. Μας είπατε ότι το 2015 πήγε καλύτερα για την ελληνική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Πριν λίγες ώρες ο κύριος Δομπρόφσκης, που δεν συνηθίζει να κάνει και πολύ θετικές δηλώσεις για την Ελλάδα, είπε ότι και το 16 πάει καλά και δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί ο περίφημος κόφτης. Και είπατε ότι και ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν τηρεί τις συμφωνίες, εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις από τις προβλέψεις και ζητά και από τους δανειστές να τηρήσουν τις δικές τους δεσμεύσεις, ιδιαίτερα για την ελάφρυση του χρέους. Κύριε Κερέ, γνωρίζετε ότι ο Αλμπέρ Καμί έχει γράψει ένα θαυμάσιο κείμενο για τον Σύσυφο. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων νιώθει ότι ζει το μύθο του Συσύφου. Γιατί εμείς εφαρμόζουμε τις μεταρρυθμίσεις, υπάρχουν θετικές προοπτικές και έρχεται ο κύριος Σόιμπλε τώρα και λέει να αναβάλουμε τα μέτρα για την ελάφρυση του χρέους γιατί εγώ σε ένα χρόνο έχω εκλογές στη Γερμανία. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς την σειρά των πραγμάτων. Από ό,τι ξέρω συζητάτε οι δανειστές με τις ελληνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα τεστ των υδάτων στα μέσα του 17 για ένα μικρό δάνειο από τις αγορές. Σας ερωτώ ποια είναι η λογική σειρά των πραγμάτων μπορεί να βγει η Ελλάδα να δανειστεί στις αγορές στα μέσα του 17 χωρίς προηγουμένως να έχει βρεθεί μια συμφωνία Διεθνές Νομεσματικού Ταμείου Κομισιών Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ESM για, για την εξειδίκευση όσον αποφάσισε το Eurogroup. Επίσης, εσείς συζητάτε ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση από τις αρχές του 2017 αν αναβληθεί ελάφρυνση του χρέου όπω θέλει ο κύριο Σόιμπλε, αν εσεί αναγκαστείτε να αναβάλλετε τη συμμετοχή τη Ελλάδα στο quantitative easing, είναι δυνατόν να προχωρήσει η εφαρμογή τη συμφωνία και να βγούμε να τεστάρουμε τι αγορέ και να πετύχει το πρόγραμμα. Και ένα τελευταίο. Διάβασα ότι την περασμένη εβδομάδα μετήχατε σε... Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Ότι μετήχατε σε μια συνάντηση κορυφαίων υπηρεσιακών παραγόντων στην Ουάσιγκτον είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη συζήτηση προέκυψε αδιέξοδο και εχθρικό κλίμα και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα ή μας ετοιμάζεται μία λύση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συμβάλλει σε αυτό. So, um, again, thank you for the... Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει αν όλα τα μέρη δεν ανταποκριθούν στις ε, υποχρεώσεις τους που είναι σαφείς. Η συμφωνία του Eurogroup του Μαΐου του 16. Εκεί αναφέρομαι. Όχι, του 16, Ναι. Δεν θα υπάρχει άλλος οδικός χάρτης. Αυτό που συμφωνήθηκε στο Eurogroup, στο Eurogroup στις 24 Μαΐου ισχύει. Διστάζω να μπω σε μια συζήτηση που είναι πολιτικής φύσεως μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και κρατών μελών σχετικά με το πώς ακριβώς και πότε θα γίνει η συζήτηση για το χρέος. Ο πρόεδρος του Eurogroup θα το οργανώσει αυτό το πράγμα και θα είναι ε, συζήτηση μεταξύ κρατών μελών. Αυτό που κάνουμε ως ένα θεσμικό όργανο είναι να προετοιμάσουμε τη συζήτηση, να προπαρασκευάσουμε δηλαδή τα πράγματα και μετά οι εκλεγμένες κυβερνήσεις θα αποφασίσουν πώς και πότε θα κάνουν τη συζήτηση αυτή. Εμείς προετοιμάζουμε το έδαφος. Αυτό που κάνουμε λοιπόν στην πράξη είναι ότι συζητούμε με τα άλλα θεσμικά όργανα, και αναφερθήκατε συζήτηση στην Washington την περασμένη εβδομάδα. Είναι μία από πολλέ τεχνικέ συζητήσει μεταξύ των τεσσάρων θεσμών. Και αν είσαστε στην αίθουσα παρόν, θα, δεν θα είσαστε τόσο ανήσυχο Κάθε εβδομάδα περίπου, κάθε δεύτερη εβδομάδα κάνουμε συναντήσει. Ε, οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να συνεδριάσουμε οι τέσσερις θεσμοί για να κάνουμε απολογισμό της κατάστασης και να δούμε τις απόψεις των ειδικών μας. Δεν υπάρχει τίποτα το θεαματικό. Καλά πήγε, ε, προετοιμάστηκαν κάποια τεχνικά θέματα. Προς το παρόν, όπως είπα, ως επιτοπλίστων, στον ESM ε εξετάζονται βραχυπρόθεσμα μέτρα, αυτή είναι η προτεραιότητα που σας απασχολεί και μετά προετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη συζήτηση. Ε, και συνεργαζόμαστε με το Δουνουτού που στα πλαίσια του άρθρου 4 τη συζήτηση με την, ε, κάνει συζήτηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το DS, ε, δηλαδή η ανάλυση για την βιωσιμότητα του χρέους. Ε, θα πρέπει να υπάρχει όμως το πλαίσιο, να γίνουν κατανοητές οι διαφορές και να προετοιμαστεί η συζήτηση. Δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο. Επαφίεται στους πολιτικούς ηγέτες το πότε θέλουν να κάνουν τη συζήτηση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η συζήτηση είναι χρήσιμη και χρειάζεται ε, για ε, όλα αυτά τα, τα, τα, θέματα που αναφέρατε. Και εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Τώρα για την ποσοτική χαλάρωση του QE. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, ΕΚΤ ήταν σαφές στις 22 Ιουνίου. Είχαμε μια δήλω... Κάναμε μια δήλωση που εξηγεί ότι θα εξετάσουμε πιθανές αγορές ελληνικών ομολόγων ε, και υπάρχει το PSPP, για το, όπως λέμε, για τα ε, ε, ελληνικά ομόλογα, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έγινε σε σχέση με την βιωσιμότητα και άλλα βέβαια θέματα αξιολόγησης κινδύνου. Και εδώ η σειρά των πραγμάτων είναι σαφής. Πρέπει να ξέρουμε περισσότερα για τα μέτρα, για το χρέος, πώς θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα πριν προχωρήσουμε στα βήματα αυτά ως Ευχαριστώ. Σβέν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τον ρόλο της ΕΚΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα ζητήματα. Στην αρχή του καλοκαιριού, πέρσι, η ΕΚΤ έθεσε ένα το στον ELA και δικαιολόγησε την απόφασή της αν και ήδη υπήρχε ένα ανώτατο όριο για τις κυβερνήσεις, το τι μπορούν να επενδύσουν δηλαδή στον τραπεζικό τομέα. Δεύτερον, η δικαιολογία ήταν ότι μπορεί να μην υπάρχουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύσεις, αν και το κούρεμα των περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών τραπεζών ήταν ε, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σε άλλα προγράμματα. Και αυτό ε, δημιουργεί ερωτήματα. Ήταν ισότιμη η μεταχείριση της Ελλάδας τα μέτρα για τον ELA, για τον περιορισμό δηλαδή του ELA στην Ελλάδα, ήταν δικαιολογημένα και αυτό επηρέασε τρομακτικά την ελληνική οικονομία. Στις 11 Νοεμβρίου επίση, 2014, η εφημερίδα New York Times δημοσίευσε δικά σα email προς τις ε, κυπριακές αρχές σχετικά με το πώς θα αξιοποιήσουν το μηχανισμό λέει, τα email τα έχετε υπογράψει εσείς. Ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε εσείς γιατί βοηθήσατε ουσιαστικά τις αρχές της Κύπρου, αλλά δεν βοηθήσατε τις ελληνικές αρχές. Είναι ισότιμη μεταχείριση αυτό των δύο χωρών. Και χθε η Επιτροπή μας αποφάσισε τα εξή. Το κείμενο λέει τονίζει τον ρόλο της ε, ΕΚΤΑ, τον Ιούνιο του 2015 όσον αφορά το γελέι στην Ελλάδα και καλεί επίσης την ε, ΕΚΤ να σχολιάσει την στάση της, την αντίστοιχη στάση της όσον αφορά το ELA για την Κύπρο. Η κατάσταση δεν είναι σαφής. Η ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε σε μια στατική και δυναμική σε αρτήσει του αποτελέσματο των ε, δοκιμών αντοχή των τραπεζών. Για να εξετάσει λέει, δηλαδή, κατά, κατά πόσον θα συνεχιστούν οι περιορισμοί στον ΙΕΛΕ ή όχι. Και υπογραμμίζει ότι η έλλειψη ασάφεια στη συμπεριφορά τη ΕΚΤ δεν αποτελεί ασφαλή δικαίου, ούτε συμβάλλει προ την σταθεροποίηση των οικονομιών. Θέλω να μου πείτε, πραγματικά, τι ρόλο διαδραμάτισε η ΕΚΤ προκειμένου. θέλουμε ακόμα καλύτερα να έχουμε όλη τη σχετική τεκμηρίωση. Αυτό που είπα, ισχύουν ή όχι. Ήταν ισότιμη μεταχείριση τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Μεταχειριστήκατε ισότιμα τι ελληνικέ τράπεζε και τι κυπριακέ. Θέλω πλήρη σαφήνεια. Πώ λειτουργεί το πλαίσιο του ELA. Θέλουμε νομική ασφάλεια όσον αφορά τη λειτουργία του ELA προς τις δύο χώρες. Ευχαριστώ για το ερώτημα, για τα ερωτήματα. Το θέμα είναι, από ό,τι κατάλαβα, ισότιμη μεταχείριση και δι Ελλάδας-Κύπρου σε όρους ε, φρεγγιότητας και ρευστότητας. Αυτές είναι οι δύο πτυχές. Όσον αφορά την παροχή ΕΛΕ στην Ελλάδα, εφαρμόσαμε ακριβώς τους ίδιους κανόνες στην περίπτωση της Ελλάδας, ό,τι κάνουμε και με τις άλλες χώρες. Και μην ξεχνάτε ότι η απόφαση περί είναι απόφαση της κρατόπους κεντρικής τράπεζας. Η τράπεζα της Ελλάδος ζητάει, εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, ΕΚΤΑ βάσει του 14.4 του καταστατικού της ε, ΕΚΤΑ ελήφθη σχετική απόφαση. Για να μην το πω ε, νομικά, το βάρος της απόδειξης είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Από εκεί πέρα είναι η κρατόπους κεντρική τράπεζα, η τράπεζα της Ελλάδος που αποφασίζει. Το πράξαμε αυτό σε διάφορες περιπτώσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα βεβαίως. Το κάνουμε στην Κύπρο όταν είχαμε στείλει και την επίσημη προειδοποίηση το 2013. Νομίζω τον 25 Φεβρουαρίου του 2013 αν δεν κάνω λάθος ήμουν στην Κύπρο λόγω της έλλειψης προγράμματος και έλλειψης χρηματοδότησης στην Κύπρο, είχαμε πει, λόγω της ε, επιδείνωσης δηλαδή της κατάστασης την εποχή εκείνη και δεδομένου του πρόβληματος της λαϊκής, η ΕΚΤ δεν θα συνέχισε την συνέχιση της παροχής ΕΛΕΗ προς τις τράπεζες της Κύπρου, εκτός αν ενισχύονταν οι τράπεζες. Άρα, πρόγραμμα. Αυτή ήταν η δημόσια ανακοίνωσή μας τότε. Και έγινε αυτό λόγω της επιδρούμενης φερεγγιότητας των τραπεζών. Η κατάσταση δεν πήγαινε καθόλου καλά στη χώρα και δυστυχώς γνωρίζετε ότι η αξιοπιστία των τραπεζών επηρεάζει και την αξιοπιστία μιας κυβέρνησης. Το κάναμε αυτό στην Κύπρο, το κάναμε πέρσι στην Ελλάδα, όπως είπατε και εσείς. Με διαφορετικούς τρόπους η κατάσταση εν γέννη ήταν διαφορετική. Πρώτον, θέσαμε ένα το όριο Μάλλον πρώτα φροντίσαμε ο ELA προ τι ελληνικέ τράπεζε να μην χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει τα ελλείμματα τη ελληνική κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση δεν είχε πρόσβαση εννοείται στην αγορά. Δεν θέλαμε λοιπόν να παρακαμφθεί ο σκοπό του ELA. Δεν θέλαμε εμέσω να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία, την ελληνική κυβέρνηση. Δεν, θέλουμε, θέλαμε να δώσουμε λεφτά δηλαδή στι τράπεζε και οι τράπεζε να χρηματοδοτήσουν τον προπολογισμό επειδή δεν υπήρχαν άλλοι πόροι. Γι' αυτό βάλαμε λοιπόν το όριο της έκθεσης των τραπεζών στην κυβέρνηση, σε δανεισμό προς την κυβέρνηση. Και όπως είπα φροντίσαμε ο ΙΕΛΕΙ να μην χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση του ελλείμματος. Μετά, αργότερα, φτάσαμε σε ένα σημείο που και πάλι, ε, όπως έγινε και στην Κύπρο το 2013, αλλά εδώ είχε μεγαλύτερε διαστάσει, δεν αφορούσε μόνο μία τράπεζα, θα μπορούσε να έχει επηρεάσει η κατάσταση όλο το τραπεζικό σύστημα. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο όπου η φερεγγιότητα και τη κυβέρνηση και των τραπεζών λόγω τη έκθεσή του ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και εμεί ε, ασχοληθήκαμε και με το θέμα τη ρευστότητα και με τι εγγύσει που μπορούσαν να παράσχουν οι τράπεζε. Τα προβλήματα αυτά ανέκυψαν όλα μαζί. Ε, προβλήματα μεγάλη έκθεση σε αβεβαιότητες. Δεν υπήρχε πολιτική λύση για την αξιοπιστία της κυβέρνησης, γι' αυτό και θέσαμε ανώτατο όριο στον ELA. Αυτό έγινε. Πάντως, οι καταστάσεις διαφέρουν. Με ρωτήσατε μετά για το τι κάνουμε εμείς με τις εθνικές αρχές, πώς μιλάμε κλπ. Έχουμε. Δεν μπορώ τώρα να σχολιάσω διαρροές εφημερίδες, αλλά αυτό που μπορώ να σας ε, πω είναι ότι βεβαίως εννοείται μιλάμε με τις ε, Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, συζητούμε την ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων, των εγγύσεων που παρέχουν. Αυτό κάνουμε ε, κάθε μέρα. Μιλάμε με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, της Τράπεζας της Κύπρου κλπ. Μιλώ με όλους τους διοικητές και φροντίζουμε τα περιουσιακά του στοιχεία, που παρέχουν είναι υψηλή ποιότητα. Εννοείται. Επίση, κινητοποιούμε δάνεια προ επιχειρήσει με τέτοια, τέτοιες εγγυήσεις για να βελτιώσουμε τη ρευστότητα στην οικονομία. Είναι και αυτό μέρος της καθημερινής μας δουλειάς. Συγγνώμη για την ισότιμη μεταχείριση όμως δεν το σχολιάσετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση, αλλά μπορείτε γραπτός να δώσετε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα σχετικά με την απομείωση του χρέου και την ισότιμη μεταχείριση. Κοιτάξτε, αν έχετε ερώτηση, ε, ευχαριστώ να απαντήσω. Δεν έχω το εγγραφό. Πρέπει να το δούμε με το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά ευχαρίστω θα το θέσω το ερώτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος. Ε, κύριο, η, η, κυρία Λούκε. Ε, θα, α, η, κυρία Καηλή. Α, όχι, κυρία Περβάνης Περάης. Στα γαλλικά να πω το δεν θέλω σχόλιο για τι αποφάσει του Eurogroup. Ίσως θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι περισσότερο το Eurogroup, αλλά αυτό που με απασχολεί είναι το εξή. Τι είναι στην Ουάσιγκτον. Φαίνεται ως προς το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ ότι το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ βλέπει το ελληνικό χρέος με τρόπο διαφορετικό από τη ευρωπαϊκή θεσμή. Το βλέπουν αλλιώ οι υπουργοί, ειδικά από ό,τι φάνηκε και στι 24 Μαου. Ποιε είναι οι διαφορέ προσέγγιση όσον αφορά το ελληνικό χρέο μεταξύ ΔΝΤ αφενό και ΕΚΤ από την άλλη. Κύριε Καηλή. Um, so thank you for your... Greece. Ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας 7 χρόνια τώρα. Η δεύτερη αξιολόγηση, αν είναι επιτυχής, θα αποτελέσει για την ΕΚΤ αρκετή πρόοδο για να μας δώσει την ποσοτική χαλάρωση. Μετά τη δεύτερη αξιολόγηση δεν θα υπάρχουν ε, οικονομικές ανάγκες για ένα χρόνο. Μπορείτε να φροντίσετε ε, ώστε η υπερφορολόγηση δεν θα συνεχιστεί και θα υπάρξουν επιστροφές. Επίσης, πιστεύετε ότι είναι η δημοσιονομική στόχοι ε, φυκτοί και η ΕΚΤ θα προβλέψει σταθερό αντικειμενόμενο επιτόκιο όπως είχαν υποσχεθεί στην προηγούμενη κυβέρνηση. Τρίτη ερώτηση δύσκολη. Η ΕΚΤ προτίθεται να συνεχίσει να αγοράζει περιφερειακά ομόλογα αν αυξηθούν τα ελλείμματα και η προοπτική είναι λιγότερο, είναι λιγότερο βιώσιμη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θα με ενδιέφερε η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα. Μιλήσατε για την κεφαλαιοποίηση που βελτιώθηκε, αλλά δεν είπατε πολλά για τις προοπτικές κερδών ε, για τις ε, τράπεζες. Αυτό σε σχέση και με την κριτική ε, για τα αρνητικά επιτόκια, η διατήρηση αποθεματικών στοιχίζει πολύ. Ε, ε, αυτή τη στιγμή δεν είναι ε, σύμφωνες οι καταθέσεις. Πώς μπορούν να κερδίσουν χρήματα οι ελληνικές τράπεζες και τι επιχειρηματικό μοντέλο έχουν οι ελληνικές τράπεζες για να εξασφαλίσουν την επίτευξη κερδών. Ευχαριστώ. Θα δώσω μια σύντομη απάντηση στις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση της κυρίας Μπερέζ για τις πιθανές... Α, θα μιλήσω γαλλικά. Η διαφορά μεταξύ της προσέγγισης ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και ευρωπαϊκών θεσμών. Πώς βλέπουν οι δύο πλευρές το χρέος. Ναι, υπάρχουν διαφορές. Άλλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο, άλλο το πλαίσιο του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ ή άλλες χώρες. Δύο είναι οι διαφορές κυρίως, οι αντικειμενικές. Πρώτον, τα δάνεια του ΕΣΜΟ, του ΕΣΜ έχουν πολύ καλύτερους όρους από τα όρια του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Εκεί το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ προκειμένου στην Ελλάδα δίνει πολύ χαμηλά δάνεια, αλλά σε συνεργασία με τον ESM. Έχουμε μετά τη διάσταση της βιωσιμότητας του χρέους και έχουμε και τις, ε, την πολιτική δέσμευση των υπουργών του Eurogroup ε, που έχουμε στην περίπτωσή μας και δεν έχει το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Δεν θα σχολιάσω το πολιτικό κομμάτι και πώς το βλέπει ενδεχομένω ε, το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Πάντως το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, αυτή είναι η θέση του, ε, δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη στους ε, υπουργούς του Eurogroup. Όμως, οτιδήποτε κάνουμε ή δεν κάνουμε, λαμβάνεται υπόψη στην μελέτη αξιολόγησης του χρέους, της βιωσιμότητας του χρέους. Και όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη στην περίπτωση μέτρων για την απομείωση του χρέους. Αυτά έτσι είναι οι βασικές διαφορές. Ε, μια ερώτηση αφορούσε την, το QE και αν ε, η επιτυχής αξιολόγηση είναι αρκετή. Είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για το QE. Για να είναι επιλέξιμες οι χώρες για αυτό το πρόγραμμα, το QE θα πρέπει να συμμορφούνται ε, προς το πρόγραμμα οικονομικής ε, στήριξης. Αυτό είναι αναγκαία συνθήκη και αποκαταστάθηκε η συμμόρφωση της Ελλάδας με βάση την πρώτη αξιολόγηση εις ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα, δηλαδή των ελληνικών ομολόγων ως εγγύηση. Γιατί υπάρχει συμμόρφωση προς το πρόγραμμα. Αλλά για την αγορά ομολόγων χρειάζεται ένα πρόσθετο επίπεδο ε, εγγυήσεων, διασφαλίσεων και σαφήνειας. Και θα πρέπει να δούμε και τα μέτρα για το χρέος. Αυτή είναι η άλλη συνθήκη. Τώρα, αν μπορεί να δώσει σταθερό επιτόκιο στην Ελλάδα. Όχι, λυπάμαι, αλλά όχι. Τα επιτόκια είναι, καθορίζονται από την αγορά. Α, και μια άλλη ερώτηση. Για τον ESM, αν μπορεί να αλλάξει το, τους όρους των δανείων. Αυτό δεν θα το σχολιάσω, γιατί είναι θέμα του ESM. Αλλά οι συνθήκες της αγοράς είναι αυτές που είναι. Και καθορίζονται από τις κεφαλαίες αγορές μπορούμε να συνεχίσουμε να αγοράζουμε περιφερικά ομόλογα αν ε, ε, ε, επιδεινωθεί η κατάσταση. Έχουμε κάποια κατόφλια, αυτό είναι σαφές και κατανοητό από όλες τις κυβερνήσεις, ότι μπορούμε να αγοράσουμε με βάση ένα συγκεκριμένο κατόφλιο ομόλογα. Αυτό δεν θα αλλάξει. Ο κύριος Λούκας για τη γερδοφορία των ομολόγων, αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα για το πρόγραμμα. Τα ελληνικά ομόλογα ανακεφαλαιοποιήθηκαν και είναι φερέγγια σε ό,τι αφορά τους ρυθμιστικούς δείκτες και ε, ε, είναι ε, φερέγγια, ακόμα και σε αρνητικό σενάριο στο stress test που κάναμε. Η κερδοφορία είναι μια πρόκληση, είναι μια πρόκληση για όλα τα ομόλογα της Ευρωζώνης άλλωστε, λόγω της δομής υψηλού κόστους, λόγω του αδύναμου ε, οικονομικού περιβάλλοντος και ελλειπούς ανάπτυξης. Αυτό ισχύει κυρίως στην Ελλάδα που έχουμε, ε, υπάρχει το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Αυτό θα το δούμε σταδιακά και θα πρέπει να ε, λειτουργήσουν τα ίδια τα ομόλογα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δράσει η κυβέρνηση εμείς. Είπαμε ότι πρέπει αυστηρά να εφαρμοστούν τα κριτήρια για τα ομόλογα, γιατί θέλαμε να υπάρχει ε, αντιστροφή των προγραμμάτων για τα ομόλογα για να τα δουν μέσα από τη δυνατότητα κερδοφορίας τους. Αρχίσαμε λοιπόν ε, ε, με την αλλαγή των ομολόγων. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε την πρωτοβουλία Τη ελληνικής κυβέρνησης ε, και μετά ο επόπτης θα κάνει τον έλεγχο. Η ΕΚΤ δεν είναι ε, υπεύθυνη για το θέμα αυτό των ομολόγων. Ε, τώρα, για τα αρνητικά επιτόκια και η πολιτική μας, βεβαίως αυτό είναι το λιγότερο πρόβλημα, το μικρότερο πρόβλημα για την Ελλάδα. Τα αρνητικά επιτόκια ε, εφαρμόζονται όταν υπάρχουν υπερβολικά ε, πλεονάσματα ε, στην ECB, στην ΕΚΤ, που αυτό δεν αφορά την Ελλάδα γενικά για την Ευρωζώνη, αυτό είναι άλλη συζήτηση. θα έλεγα όμως ότι τα αρνητικά επιτόκια μέχρι τώρα αντιμετωπίστηκαν θετικά από τα ευρωπαϊκά ομόλογα γιατί στηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία και συμβάλλουν στην μείωση των ε, ε, απολειών ε, από δάνεια. Όπως είπαμε πολλές φορές, αυτό θα το δούμε. Θα δούμε δηλαδή τα χαμηλά επιτόκια και τα αρνητικά επιτόκια. Αυτό κάποια στιγμή θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα την κερδοφορία των ομολόγων, αλλά όπως σας είπα, στην Ελλάδα αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα με τα ομόλογα. Αν η κερδοφορία είναι χαμηλή, είναι χαμηλή γενικότερα στην Ευρωζώνη, γιατί ε, το, τα κόστη είναι πολύ υψηλά σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Ε, υπάρχει δηλαδή ανάγκη ε, εξυγίανσης εδώ στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Αυτό όμως είναι αντικείμενο άλλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας και προφανώς θα συνεχίσουμε να είμαστε σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εν και γενικότερα στα πλαίσια του νομισματικού διαλόγου. Ευχαριστώ.